όπου ε, υπάρχουν περισσότερες παραβιάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα είναι οι συζητήσεις ε, για περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και περνάμε στην Ρουάντα. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Κοράο πρώτα. Thank